Okay, colleagues, if everyone could start taking their seats. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Θα ήθελα να καθίσουμε σας παρακαλώ. Thank you, colleagues. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ πίσω στην αίθουσα είτε να καθίσετε είτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Δεν θα, είναι, δεν θα χρειαστούμε ιδιαίτερο χρόνο, αλλά χρειαζόμαστε ησυχία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε και εσείς ε, συνάδελφοι, εδώ είμαστε τρεις επιτροπές, προϋπολογισμός, ε, ΑΦΕΤ και ΔΕΒΕ. Ε, έχουμε εδώ λοιπόν εμένα ως πρόεδρο και δύο ανταπρόεδρους δίπλα μου και έχουμε σκοπό την ψήφιση του κειμένου που μας αφορά και να σας πω πως καταρχήν πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και το μοναδικό σημείο είναι το 4 Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δημιουργία Εγγυήσεων έγκριση αυτού. Αυτό θα ψηφίσουμε. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Το μόνο που θα σας πω είναι πως έχουμε εδώ μια προσωρινή συμφωνία που αν ε, ψηφιστεί, υπερψηφιστεί σήμερα, θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια με διαδικασία fast track την Δετάρτη το απόγευμα. Αυτό έχουν συμφωνήσει οι τρεις ε, εισηγητές από τις τρεις ε, επιτροπές και τις αντίστοιχες πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι εδώ ε, η Αντιπροεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμού θέλει να πει δύο λόγια. Ναι, παρακαλώ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να ζητήσω, ε, να, να παρουσιάσω, με συγχωρείτε, την ε, Ε, να σα ε, πω πω ο πρόεδρο μα, κύριο Σορβί, δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ε, λυπάται πολύ. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ τη σημασία που έχει το κείμενο αυτό. Γιατί τα όσα κάνουμε σήμερα εδώ είναι σημαντικά. Και θα τονίσω το εξή. Καταρχήν, υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία πολιτών στην Ευρώπη που θέλουν εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να μείνει στη χώρα του και να ε, βοηθήσουμε επίσης και τις χώρες transit, οπότε ό,τι και να κάνουμε χρειάζεται να ε, συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό που μας ζητάει ο κόσμος. Ωραία λοιπόν. Ε, επειδή λοιπόν δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα συνεχίσουμε. Σας ζητώ να περάσουμε στο 3, έγκριση των πρακτικών. Έχουμε τα πρακτικά των κοινών συνεδριάσεων τη 11 η Απριλίου του 2017. Αν έχετε σχόλια σας παρακαλώ προς τη γραμματεία, διαφορετικά θεωρούμε πως έχουν εγκριθεί και μπορούμε να περάσουμε στο 4 που είναι η ψηφοφορία πριν ψηφίσουμε Έχουμε ένα ιστορικό κείμενο, εμπλέκει τρεις ε, επιτροπές, τρεις συζητητές και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Κούκαν, για παράδειγμα, να μας πει δύο λόγια από την ΑΦΕΤ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως το θέμα αυτό χρειαστήκε χρόνο ρεκόρ για να φτάσει μπροστά σας. Οι τρεις εισηγητές χρειάστηκε με ε, πολύ ιδιαίτερο τρόπο να το συμφωνήσουν ε, με όλες τις συζητήσεις που έγιναν και σε όλες του τις ε, πτυχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους μας βοήθησαν. Θα ήθελα την κυρία Γκαρδιάς... Ζάμπα Λουρμπιάλ και τον κύριο Φρουντζούλικα να τους ευχαριστήσω ως συνεισηγητές ιδιαίτερα και να σας πω πώς αποδεικνύει ε, τούτη η συμφωνία πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τόσο ακαθόδες θέμα με έναν τρόπο που κατάφερε ε, να συνδυάσει όλα τα συμφέροντα τα οποία ε, εδώ εμπλέκονται και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν. τώρα ο κύριος Φρουντσούλικα από την Επιτροπή Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους άλλους ε, συνεισηγητές, την κυρία Κουαρδία Σάπαλ και τον κύριο Κούκαν, όπως επίσης και τους Κιώδης, ε, το προσωπικό μας συνεργάστηκαν εξαιρετικά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις Προεδρίες των Τριών Επιτροπών, τους συντονιστές, να σας πω πως συνεργαστήκαμε και χρειαστήκαμε να ακολουθήσουμε μια δύσκολη διαπραγματευτική διαδικασία και ήταν πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα επικοδομητικό το ότι καταφέραμε να στηρίξουμε ε, αλλήλους και να παρουσιάσουμε μια στέρεη θέση εμείς ως θέση του Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά το τελικό κείμενο θα το υπερψηφίσω. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κινητοποιήσει μέχρι 44 δις σε επενδύσεις και αυτά για βιώσιμη ε, και κοινωνική ανάπτυξη έτσι ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές οι χώρες εταίρες στην Αφρική και στην ε, Ανατολική γειτονία της Αυρωπαϊκής ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θα εστιάσουμε περισσότερο στι γυναίκε, στα παιδιά, στη, θέση, στη δημιουργία θέσεων εργασία και ε, στα όσα αφορούν τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει και να σα πω πω η εφαρμογή αυτού του Ταμείου δεν θα είναι εύκολη, αλλά μέσω τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, στο Στρατηγικό Συμβούλιο ως παρατηρητή, μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, θα τα καταφέρουμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις αρμοδιότητές μας έτσι ώστε να εξετάσουμε αυτό το εργαλείο και να είμαστε σίγουροι πως το ΕΤΒΑ θα ανταποκριθεί ε, στους στόχους του. Είμαι σίγουρος πως θα αποτελέσει πολύ πετυχημένο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προωθήσει τις αξίες μας και σίγουρα πιστεύω πως το καλύτερο είναι όλοι μας να το υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ και τελευταία η κυρία Γκαρδιά Σάβαλ από την Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή θέλουμε να ψηφίσουμε. Ανυπομονούμε. Οπότε με μία φράση να σας πω το εξή. Εμείς βελτιώσαμε τους στόχους αυτού του Ταμείου και μάλιστα οι βελτιώσεις είναι σημαντικές και σε επίπεδο σχεδιασμού. Οπότε ας υπερψηφίσουμε. Και λίγες ευχαριστίες απλώς και στους δύο συνεισηγητές γιατί πιστεύω πως συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά στις τρεις επιτροπές. Η συνεργασία αυτή ήταν θετική και μάθαμε πώς μπορούμε να το κάνουμε με τρεις διαφορετικές επιτροπές και θα ήθελα να το επαναλάβω. Η γραμματεία των τριών επιτροπών επίσης μας υποστήριξε πολύ σημαντικά γιατί αν πάντα η συνεργασία της γραμματείας είναι σημαντική το γεγονός πως μας συντόνισε και ήμασταν τρεις διαφορετικές επιτροπές ε, ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε σε όλους τους Τεχνικού τριμερεί διαλόγου, στου οποίου συμμετείχαν εργαζόμενοι για ώρε, ε, πρέπει να σα πω ότι έτσι μετά του τεχνικού τριμερεί διαλόγου, καταφέραμε εμεί του πολιτικού τριμερεί διαλόγου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέσα σε τέσσερι ε, με ε, τέσσερις μήνες και μετά από 60 ώρες διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους και κυρίως και τη γραμματεία της δικής μου πολιτικής ομάδας, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ωραία λοιπόν. Θα ψηφίσουμε το πακέτο με μιας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξέρω ποιοι δεν έχουν κάρτες, οπότε θα σας προσθέσω. Μου έχετε δώσει τα ονόματά σας. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε πρόβλημα τεχνικό γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω να αλλάζουν και τα νούμερα. Λοιπόν, ξανά. Με συγχωρείτε συνάδελφοι. Γιατί ξαφνικά πέσαμε στους 75, οπότε... Ξέρω πως κάποιοι δεν έχετε κάρτα, αλλά σας παρακαλώ πολύ δώστε μου το όνομά σας για να σας προσθέσουμε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε ψηφίσει όλοι. Πέρας. 76 υπέρ, 10 κατά, 3 αποχές. Δεν θα το ελέγξουμε, νομίζω κύριε Πρέντετα, είναι πολύ ε, σαφές το αποτέλεσμα. Ωραία, ονομαστική λοιπόν, είναι ονομαστική η ψηφοφορία, σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ και όλο το προσωπικό που κάνει καταπληκτική δουλειά και όλους τους ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης αρχίζει στις 8 ακριβώς, εδώ.